Ε, καλό σας απόγευμα. Να ενημερώσω το σώμα ότι ε, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 δεν υπάρχει αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία κανένα διορθωτικό από αυτά που ανακοινώθηκαν χθε στις 5. Τα διορθωτικά θεωρούνται εγκεκριμένα λοιπόν. Και τώρα προχωρούμε στην